Άδελφοι. Καλημέρα. Παρακαλώ καθίστε. Όπως ξέρετε είναι μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και φορολογικών ε, υποθέσεων. Ε, Καλώς ορίζω τον συνάδελφο κύριο Γέζεκ ε, και τον Επίτροπο Μοσκοβισή, τον αρμόδιο Επίτροπο για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνία. Αυτό μας απασχολεί σήμερα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ επίκαιρη συζήτηση γιατί την προηγούμενη εβδομάδα όπως όλοι ξέρουμε ο κύριος Μοσκοβισή παρουσίασε μια πρόταση για δίκαιη φορολογία για την ψηφιακή οικονομία και βεβαίως ε, δεν θα σας προξενήσει εντύπωση το ότι η πρόταση αυτή ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος την Επιτροπή μας όπως ξέρετε μόλις έγκριναμε, ε, ψηφίσαμε την ε, διαδικασία διαβούλευση στην, ε, στην οδηγία για την κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων και από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση σύγκλησης ε, μακροπρόθεσμη κατόπιν όπως ξέρετε η Κομισιόν ε, εισήγαγε μια βραχυπρόθεσμη λύση με αυτό το 3% το οποίο αποτελεί μια Και για μας βεβαίως πάντα η καλύτερη λύση είναι να φορολογήσουμε τα κέρδη, αλλά γεγονός είναι ότι το να πιέζουμε βράχη πρόθεσμα για αυτήν την ε, λύση θα είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Προσωπικά λοιπόν καλωσορίζω το πακέτο αυτό ε, και επιπλέον ε, ο Επίτροπος Μοσκοβισή έχει υποβάλει συνολικά έξι νομοθετικές προτάσεις για το σύστημα ΦΠΑ σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ και έχουμε ήδη προχωρήσει σε δύο από αυτές τις προτάσεις και οι συγητές μας ξεκίνησαν ε, τις προτάσεις ε, επί των λοιπόν νομοθετημάτων. Έχουμε λοιπόν και την πρόταση για ένα οριστικό καθεστώς που αναμένουμε και αναμένουμε ακριβώ ε, το τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Όπως βλέπετε εμείς είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε γρήγορα στην ΕΚΟΝ και τώρα δίνω τον λόγο στον Συμπρόεδρο, τον κύριο Γέζεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ρομπέρτο, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η παρουσία σας σήμερα είναι πάρα πολύ συμβολική. Έχουμε την πρώτη κοινή συνεδρίαση των επιτροπών μας και οι ε, υπηρεσίες σας έχουν παρουσιάσει διάφορες ε, πρωτοβουλίες ε, στου τομείς που μας ενδιαφέρουν και η κοινή μας συνεδρίαση είναι σημαντική όχι μόνο γιατί οι δύο επιτροπές έχουν πολλά μέλη κοινά αλλά γιατί έχουμε και κάποιες πρωτοβουλίες ε, στο μέτωπο της ε, νομοθεσίας. Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστεί η Επιτροπή μας ε, μαζί σας στενά, όπως έγινε και με τις προηγούμενες επιτροπές, τάξη 1, 2 και πάνω. Και έχουμε ακριβώς τα ζητήματα των επιβλαβών φορολογικών μέτρων, των προνομίων, την ε, διάσταση των τρίτων χωρών στην φοροαποφυγή και την απάτη του ΦΠΑ. Επίσης, ε, προσφάτως περιλάβατε για πρώτη φορά τις ε, παρατηρήσεις για τις πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στα κράτη-μέλη στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Προφανώς μας ενδιαφέρει αυτό και βεβαίως ε, κυρίως ε, του εάν ε, θα υπάρξει συνέχεια στις συστάσεις αναχώρα. Επίσης, αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στις, εξερε... στις εξελίξεις όσον αφορά τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων τρίτων χωρών του Συμβουλίου, ιδιαίτερος στο θέμα της διαφάνειας της διαδικασίας. Τέλος, θέλουμε να μάθουμε το τι έγινε με την διαδικασία επί παραβάση που κίνησε η Κομισιόν κατά κάποιων κρατών μελών μετά από τις αποκαλύψεις για τα Paradise Papers και την εφαρμογή της οδηγίας ΦΠΑ. Πριν ε, σας δώσω τον λόγο, να εξηγήσω το τι θα κάνουμε. Μετά από τις αρχικές παρατηρήσεις του Επιτρόπου, σας παρακαλώ περιοριστείτε σε 10-15 λεπτά έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Αυτή τη φορά έχουμε μείνει λίγο πίσω, οπότε θα έχουμε μόνο τέσσερα λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις, οπότε παρακαλώ να περιοριστείτε σε λιγότερο από ένα λεπτό για να μπορεί να απαντήσει ο Επιτροπός. Για να απομείνει χρόνος. Βεβαίως, Έχετε δικαίωμα να κάνετε και άλλη ερώτηση. Στον ε, πρώτο γύρο ερωτήσεων κάθε πολιτική ομάδα θα κάνει από μία ερώτηση και μετά θα περάσουμε στο σύστημα DEONT. Εάν υπάρχει χρόνος ε, θα δοθεί ο περισσότερος χρόνος στην βάση του συστήματος Και μετά θα ξαναδώσουμε τον, την Προεδρία στον Πρόεδρο της ΕΚΟΝ. Κύριε Επιτροπέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να συνεργαστώ με τη νέα Επιτροπή και την Ειδική Επιτροπή ΤΑΞ 3. Καταρχήν ε, συγχαρητήρια για τους προέδρους ε, και αντιπροέδρους για τις εκλογές τους. Καταρχήν θα ήθελα να σας εκφράσω την πλήρη ε, θέλησή μου καθώς και των συνεργατών μου. Είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Οι στόχοι, οι δικοί μας και οι δικοί σας είναι οι ίδιοι. Η πολιτική πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζεται έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να σταματήσουν οι καταχρηστικές αυτές φορολογικές πρακτικές, αλλά και οι απαράδεκτες δολοφονίες δημοσιογράφων, δημοσιογράφων οι οποίοι διερευνούν τις υποθέσεις αυτές. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες θέλετε να υιοθετηθούν, αυτές βεβαίως είναι απαραίτητες. Γιατί πρώτον το ζητούν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον ανοιχτό, χωρίς ε, εμπόδια και προσκόμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και να προσελκύσει επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω και θα πρέπει να υιοθετήσει φορολογικούς κανόνες και προδιαγραφές οι οποίες να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα. Θα μπορούσα να ξεκινήσω και από το σημαντικότερο που είναι οι προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών ήρθε η ώρα η Ευρώπη πραγματικά να αποδείξει με αποτελεσματικό τρόπο ότι θέλει να αλλάξουν τα πράγματα και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει με συνένεση. Είναι καθοριστικό και για την οικονομική μας πολιτική αλλά και για την ευρωπαϊκή εικόνα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια συλλογική, κοινή στρατηγική. Ακούω ότι Βεβαίως, όσον αφορά την CCTV, τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την φορολογική τους πολιτική, την φορολογική τους κυριαρχία. Ναι, το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να δεχθούμε εδώ ε, ο καθένας να δράμε μονομένα γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι και οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πληγούν και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υιοθετήσουμε συλλογική στρατηγική. Σε μία αντίθετη περίπτωση, αν δεν τα καταφέρουμε, οι μόνοι που τελικά θα βρεθούν κερδισμένοι θα είναι οι πολυεθνικές και οι τεράστιοι όμιλοι. Το λέω με ισχύ εδώ ενώπιον σας. Δεν είναι δυνατόν πλέον να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε το dumping, το φορολογικό dumping. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η συλλογική στρατηγική, την οποία στηρίζουμε, την οποία θέλουμε να προωθήσουμε, να προωθηθεί βάση προτεραιοτήτων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μη νομοθετικά εργαλεία που διαθέτουμε για να προχωρήσουμε προς αυτήν την πιο συνεκτική, πιο συλλογική, φορολογική, στρατηγική και πολιτική και βεβαίως ε, δεν θα αναφερθώ μόνο στους φορολογικούς παραδείσους, αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που συνεχίζει να υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να δούμε τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να συσφίξουμε τους δεσμούς μας έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να υιοθετούν ε, αυτές τις πρακτικές να μην μπορέσουν να δράσουν. Πριν από πολύ ε, λίγους μήνες ξεκινήσαμε με τον εντοπισμό αυτών των σχεδιασμών οι οποίοι έχουν σαν σκοπό να αποφευχθεί η δίκαιη φορολόγηση. Θα πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι αισιώ σε όλες αυτές οι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις να υλοποιηθούν. Αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, η οποία αφορά όχι μόνο το άξις, αλλά και την φορολόγηση των επιχειρήσεων που δρούν στον ψηφιακό τομέα, αλλά και την υιοθέτηση ενός ε, σύγχρονου συστήματος ΦΠΑ αποτελεσματικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε τις προτάσεις που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στον ε, ψηφιακό κόσμο. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ισότητα μεταξύ των φορολογούμενων αλλά και τις εξελίξεις που σήμερα παρατηρούμε στον ψηφιακό κόσμο. Σήμερα, όπως ξέρετε, η φορολόγηση των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό είναι της τάξης του 9,5% κατά μέσο όρο σε σχέση με το μέσο όρο που ισχύει στους άλλους τομείς της οικονομίας που ξεπερνάει το 23,2%. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πιο ίση μεταχείριση των τομέων της οικονομίας μας. Γι' αυτό και πρότεινα το τάξης την πρόταση αυτή η οποία ουσιαστικά προτείνει η φορολογία των επιχειρήσεων αυτών που δεν έχουν σταθερή παρουσία. Όπως ξέρετε η φορολογία ουσιαστικά βασίζεται στην φορολογική έδρα και στην σταθερότητα αυτής. Προτείνω λοιπόν να υπάρξει μια πιο ίση αντιμετώπιση αυτών των δύο διαφορετικών ε, ειδών επιχειρήσεων. Επίσης όσον αφορά τον κατακαιρματισμό, την προσέγγιση patchwork όπως τη λέμε έναν ακόμα τρόπο να υπάρξει φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Η δημιουργία αξίας θα πρέπει να υπολογίζεται με έναν τρόπο πιο ολοκληρωμένο και βλέπουμε ότι επιχειρήσει επιχειρήσεις όπως η Google, η Facebook δημιουργούν πλατφόρμες, ενδιάμεσες πλατφόρμες και θα δώσω και άλλα παραδείγματα οικονομικών πρακτικών όπως αυτές που εθωτούν η Uber και η Airbnb. Εδώ θα πρέπει να βρεθεί τρόπος δίκαιης αντιμετώπισης αυτών των οικονομικών μοντέλων. Το θέμα του ΦΠΑ. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε έναν τρόπο φορολόγησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις αυτές που δρούν κατακαιρματισμένα και οι οποίες σήμερα υποφελούνται από το εξαιρετικά κατακαιρματισμένο τρόπο φορολόγησης και πιστεύουμε ότι το διαφυγόν κέρδος ξεπερνάει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες βεβαίως για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2017, θα πρέπει να βοηθήσουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει αυτό το διαφυγόν κέρδος που επαναλαμβάνω ξεπερνάει τα 150, 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε όλους τους τομείς της οικονομίας αν κοιτάξει κανείς ε, τα συστήματα ΦΠΑ είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε όλες αυτές τις δυνατότητες φορολόγησης με ένα σύγχρονο τρόπο, με ένα τρόπο που ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα του 21ου αιώνα, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας, και βεβαίως η καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φορολογικής απάπης δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις ε, συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Έχουμε και έξω νομοθετικά ε, εργαλεία, γι' αυτό και στις αρχές του μήνα έστειλα επιστολές στη Μάλτα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ε, υποθέσεις που αφορούν τον ΦΠΑ, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βεβαίω η Επιτροπή ΤΑΞ 3 δεν θα περιοριστεί μόνο στις υποθέσεις ΦΠΑ. Είναι επίσης ε, το θέμα των φορολογικών ε, παραδείσων και χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των ε, κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικά προχωρήσει και χαιρετίζω αυτήν την προσπάθεια η οποία για πρώτη φορά έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ σημαντικές ε, επιτυχίες. Πάνω από 61 χώρες οι οποίες ε, βρίσκονταν σε αυτό το κατάλογο έχουν επιτελέσει πάρα πολύ σημαντική ε, πρόοδο. Οι 31 από αυτές έχουν δημοσιεύσει τις δεσμεύσεις τους. 28 από αυτές έχουν δημοσιεύσει και 5 δεν μας έχουν ακόμα απαντήσει. Οι 29 έχουν δημοσιεύσει μερικά στοιχεία. Τέσσερις αρνούνται να δώσουν το οποιοδήποτε στοιχείο. Η πρόοδος πάντως είναι σημαντική, η στόχη μας φιλόδοξη και εδώ και ε, αρκετούς μήνες προσπαθούμε να δικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας και τις πιέσεις μας. Δεν είμαστε όμως αφελείς. Δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει έντονη, αν θέλετε, συζήτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Αλλά θα είμαι σαφής, δεν υπάρχει σήμερα φορολογική παράδεισ, φορολογικός παράδεισος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί όμως κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχουν φορολογικές πρακτικές, επιθετικοί φορολογικοί σχεδιασμοί που έχουν σαν σκοπό την ε, μερική φοροαποφυγή. Έχουμε ακούσει εξαιρετικά ανησυχητικές παρατηρήσεις. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διάλογο με κάποια κράτη-μέλη και φυσικά είναι διατεθειμένη να συνοδεύσει τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να μεταρρυθμίσουν τις πρακτικές τους. Δεν θέλω εδώ να πω ότι τα πετύχαμε όλα, ούτε να καταδικάσω με τρόπο αμήλικτο κάποια κράτη-μέλη. Χρειάζονται προσπάθειες και θα πρέπει να τροποποιηθούν κάποιες γνωστές νομοθετικές πρακτικές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται ούτε στους ηθικούς ε, ούτε στους ε, κανόνες τους οποίους έχουμε υιοθετήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοκληρώνω και θα ήθελα να σας πω ότι δεν μπορούμε από τη μία να μιλούμε για την σύγκληση των οικονομιών μας και από την άλλη να έχουμε έναν άκρατο φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φορολογικό dumping θα μας οδηγήσει όλους στο αδιέξοδο και θα πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε μια πραγματική φορολογική σύγκληση, η οποία δεν θα είναι ποτέ πλήρης εάν δεν υιοθετηθεί το άξις και το σύστημα ευρωπαϊκού ΦΠΑ. Με την πλήρη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΕΚΟΝ και της ΤΑΞ 3 μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας πριν το τέλος της θητείας της Επιτροπής. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει πριν το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν υιοθετηθεί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είμαι δεσμευμένος και ότι θα βρίσκομαι στο πλευρό σας με όλα τα μέτρα που διαθέτω. Κάθε φορά που έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνω ότι διαπιστώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση πως παρόλες τις διαφορετικές πολιτικές σας ευαισθησίες και προσεγγίσεις, είμαστε όλοι στο ίδιο πλευρό, στο ίδιο μέτωπο. Και έχουμε όλοι δεσμευθεί, και εδώ επαναλαμβάνω την πολιτική μας βούληση, να σπρώξουμε, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. Μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας σας, μέχρι την τελευταία μέρα θα είμαστε στο ίδιο πλευρό σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοσκοβισή, λέει ο Πρόεδρος Γκολτιέρη. Και εμείς σας υποσχόμαστε ταχαίως να ενεργήσουμε όσον αφορά τη νέα δεσμή μέτρων και στις προθέσεις μας. Όντως είναι να γίνει η ψήφιση των προτάσεων μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, όντως ώστε να βοηθήσουμε και τα μέτρα αυτά να ε, θεσπιστούν, να τεθούν σε ισχύ. Και τώρα αρχίζουμε τις ε, παρεμβάσεις και ο πρώτος ομιλητής ε, είναι ο Λέντα Μασούρ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι με μεγάλη χαρά ακούσαμε αυτά που μας είπατε και ιδιαίτερα στις προτάσεις της προηγούμενης εβδομάδας που έκανε η Επιτροπή. Αναφερθήκατε στην λύση την μακροπρόθεση που είναι η φορολογία για τον τομέα της ψηφιακής ε, οικονομίας στα ίδια επίπεδα με όλους τους άλλους ε, τομείς της οικονομίας. Εδώ υιοθετήσατε 100% την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή που υιοθετήσαμε με μεγάλη πλειοψηφία πριν από 15 μέρες. δεν θέλω εδώ να σας εκφράσω και μία ε, ανησυχία μας. Η CCCTB είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο. Εδώ και μήνες το έχετε υποβάλει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Υπάρχει μία ομάδα που εδώ και 18 μήνες έχει απλώς ασχοληθεί με το πρώτο κείμενο, το CCTV. Αργούν, κολυσιεργούν. Αυτοί που είναι αντίθετοι δεν λένε τίποτα. Αυτοί που δεν ξέρουν αν θα προχωρήσει το κείμενο επίσης σιωπούν. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία κρατών μέλων που είναι η χώρα από την οποία προέρχεστε και εσύ και εγώ, οι οποίοι εξετάζουν άρθρο προς άρθρο το κείμενο αυτό και προσπαθούν να αδειάσουν το κείμενο από κάθε ουσία, από το πραγματικό του περιεχόμενο. Γι' αυτό και κάνω την ερώτηση αυτή και γι' αυτό και ανησυχώ, κύριε Πίτροπε, Πιστεύετε ότι το σύστημα είναι πιο σημαντικό από τις ε, ενδιάμεσες λύσεις και πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να οδηγηθούμε ταυτόχρονα όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ βλέπουμε ότι τα κράτη δεν φαίνεται να θέλουν να λάβουν υπόψη τους σοβαρά το θέμα αυτό και να δώσουν τις σωστές οδηγίες στους υπαλλήλους τους ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ως συνήθως συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις του Αλάν Λαμασούρ. Όντως, είναι λογικό ο, ο τύπος να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον ε, προσωρινό φόρο του 3%. Είναι κάτι το θεαματικό και γι' αυτό και ασχολήθηκα με αυτό. Αλλά εννοείται ότι το πιο σημαντικό είναι το μακροπρόθερο σχέδιό μας, το μόνιμο και τελικό σχέδιο το οποίο προσπαθούμε, στο οποίο προσπαθούμε να φτάσουμε. Σήμερα όμως υπάρχει ένα τεράστιο νομικό κενό και βεβαίως βλέπουμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις του ψηφιακού τομέα συνεισφέρουν με ελάχιστα ποσά στα ταμεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν είναι το νομικό κενό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Εγώ όμως είμαι αισιόδοξο, κύριε Βλεφτά, το γνωρίζετε και γι' αυτό και χαίρομαι γιατί βλέπω να κινούνται τα πράγματα. Έχετε όμως δίκιο πρέπει να πιέσουμε και εγώ θα το κάνω έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες αυτής της Επιτροπής. Είτε πρόκειται για το άξις, είτε πρόκειται για τη βραχυπρόθεσμη φορολόγηση. Στις δύο περιπτώσεις αυτές πρέπει να βιαστούμε. Η Προεδρία της Βουλγαρίας και της Αυστρίας είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να επιτύχουν τα πιο σημαντικά βήματα. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι θα πρέπει να κινηθούμε. Εγώ θεωρώ ότι η Προεδρία, η παρούσα, είναι μάλλον θετικά προσκύμενη και μπορώ να κινήσει κάποια θέματα σε υπουργικό επίπεδο. Mm-hmm. Να το δούμε, λέει ο Πρόεδρος και δίνει στον κύριο Κόφου το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μοσκοβίση. Και εγώ έλεγα ότι αυτή η Ειδική Επιτροπή περιμένει πώς και πώς αν μπορούμε να συνεργαστεί μαζί σας, να δώσουμε τον αγώνα για την διαφάνεια, για αποτελεσματικό φορολογικό δίκαιο στην Ένωση. Όσον αφορά την διαφάνεια, ένα θέμα που πρέπει να σας αναφέρω είναι ότι έχουμε αυτού του είδους τις εκθέσεις αναχώρα. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα πρέπει να το κλείσουμε το συντομότερο δυνατόν. Για πετε μας, κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα όσον αφορά τις μη συνεργαζόμενες χώρες που καλά τα είπατε, είναι σημαντικό, Επίτροπε, βεβαίω και δίνουμε τη μάχη για τη διαφάνεια και θέλουμε επίσης να δούμε κάποια κριτήρια τα οποία να είναι αξιόπιστα για όλο τον κόσμο. Ποια πέστε μας και σε αυτό το μέτωπο κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, μας ε, αναφέρατε για αυτό το πρόσφατο ρεπορτάζ όσον αφορά την έκθεση αναχώρα για τα κριτήρια της φορολόγησης, για τις επιθετικές ε, τακτικές και ότι εννέα χώρες έχουν τέτοιου είδους φορολογικές ε, πολιτικές και τακτικές. Τώρα τι γίνεται με το μη νομοθετικό ε, με τη μη νομοθετική επιλογή, αλλά χρειάζεται και νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιθετικές πρακτικές σε αυτές τις εννέα χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβληματιστεί για το τι θα κάνει όσον αφορά ε, την φορολόγηση των επιχειρήσεων, ε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει και πολλά πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Κοφόντου. Ξέρω κύριε Κοφόντου πόσο εσείς ε, ε, ενδιαφέρεστε για την διαφάνεια και τα τελευταία χρόνια χέρι-χέρι προχωρούν προς τα κοινέα ναι, όσον αφορά τις εκθέσεις αναχώρα δεν, έχουν, ε, δεν έχει τίποτα εγκριθεί τίποτε σε επίσημο επίπεδο και αυτό εν μέρει γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τη νομική βάση. Άλλα λέει η νομική υπηρεσία, άλλα λέει το Συμβούλιο, αλλά ναι, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτή την υπόθεση και εσείς μαζί με εμάς θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη. Μην το ξεχνάτε και εμεί ενδιαφέρομαστε για το θέμα των εκθέσεων. Αναφορά τώρα όσον αφορά τη διαφάνεια. Πρώτον, όπως ξέρετε, τη σχετική λίστα δεν την καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τα κράτη-μέλη. Αλλά στο Συμβούλιο πιέζουμε ούτως ώστε οι δεσμεύσει των κρατών μελών για τη λίστα να δημοσιοποιηθούν προς τα εκεί θέλουμε να πιέσουμε να υπάρχει δηλαδή απόλυτη διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης καθεντήρες γραμμές τις έχουμε εγκρίνει σε σχέση με τον προϋπολογισμό αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν το ίδιο. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα για τον κώδικα διοντολογίας, υπάρχει φυσικά συνεργασία και θα σας ενημερώνουμε. Τέλος, όσον αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, νομίζω ότι θα πρέπει οι χώρες να προσαρμόσουν το φορολογικό τους δίκαιο για αυτό τον διάλογο μιλούσα. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Γκουαλτιέρι. Κορβόν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Για όσο μας είπατε όσον αφορά τη φορολογική πολιτική. Από πλάσα επιχειρήσεων στη Φιλανδία έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές επικρίσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο στη Φιλανδία αυτό, όπως είπατε και πριν, ότι τα, τα κοινά πρότυπα τίθενται ένα αμφιβόλο τώρα. Είπατε και για τη φορολόγηση του παθητικού. Έχουμε έτσι αύξηση της φορολογίας, επομένως. Η αξία διαμορφώνεται από την αγορά. Και πολλές φιλανδικές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα στην Φιλανδία Γιατί πάρα πολλά καθορίζονται εκτός της χώρας μας. Άρα χρειάζεται διεθνής συνεργασία και φορολογική βάση να μετακινηθεί, να μετατοπιστεί στις χώρες τις πιο μεγάλες με περισσότερο πληθυσμό. Ας αναζητήσουμε βέβαια και κάποιες ε, θετικές απόψεις για όλα αυτά που αναπτύσσετε εσείς. Οπότε πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε δυναμικοί και αποτελεσματικοί. Πάντως, να μην σκοτώσει θεραπεία τον ασθενή. Εσείς τι θα κάνετε για όλες αυτές τις επικρίσεις, τις πολύ πρόσφατες που προέρχονται από τη Φιλανδία. Μοσκοβίση, σας ευχαριστώ πρώτα-πρώτα να σας αναφέρω ότι προσπαθούμε προς αυτό το μέτωπο για να δούμε τι θα γίνει σε διεθνή κλίμακα. Παγκόσμια τα προβλήματα, άρα εκεί θα αναζητηθεί η λύση. Οπότε και στον ΟΣΑ και στο G20 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δραστήρια. Βέβαια έχουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εσωτερική αγορά και σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να δούμε το τι σημαίνει αυτή η κατάτμιση, η διαφοροποιημένη προσέγγιση. Όλα αυτά είναι αρνητικά. Οπότε θα πρέπει αναχώρα να δούμε τις επιπτώσεις και ένα κλάδο. Προς τα εκεί. Ε, αυτή την, την κατεύθυνση έχουν οι προσπαθείς μου για το άξις. Και στο Κοινοβούλιο συμφωνείτε με αυτές τις προσπαθίες μας μεγάλη πλειοψηφία για αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε τελικά να έχουμε κοινή προσέγγιση για την απάτη, για την φοροδιαφυγή και τα να αποτελεί κίνητρο προς επένδυση η φορολογική μας πολιτική. Για το παγκόσμιο εμπόριο, για την παγκοσμιοποίηση, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό θεωρώ ότι το άξις είναι μία μεταρρύθμιση που θα πρέπει να μας βοηθήσει στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να το δούμε με ένα πνεύμα συλλογικό και αθετικό Βίρνικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μία σειρά ερωτήσεων κύριε Επίτροπη για το CCTV. Νομίζω ότι Άννα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση των μεταρρυθμίσεων για τις άλλες επίρρες δηλαδή. Ποιο θα είναι το τίμημα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φορολογικού στις ΗΠΑ. Τι θα γίνει με το CCTV σε σχέση με αυτή τη μεταρρύθμιση τώρα όσον αφορά τα μεταβατικά διάμεσα μετρονομίζετε ότι υπάρχει ένας ε, κίνδυνος αυτά να προσδεθούν στη δικαιοσύνη. Ε, ότι δηλαδή είναι παράνομο για συγκεκριμένε εταιρείε. Επίση, πώς θα αποφύγετε το πώς δεν θα μετακυληθούν αυτοί οι φόροι στον καταναλωτή και πώς θα αποφύγουμε τη διπλή φορολόγηση. Πώς επίσης θα αναγκάσετε ε, κάποιες ε, εταιρείε να πληρώσουν του φόρους ενώ δεν έχουν έδρα εδώ. Στην πρόταση αυτή μεταρρύθμιση για το, την εταιρική φορολόγηση θα πρέπει να δούμε πού είναι ο χρήστης και πού είναι πού δημιουργήθηκε το κέρδος. Επομένως, θα πρέπει από κάθε χρήστη να έχουμε τη σχετική πληροφορία, σεβόμενη βέβαια και τον ιδιωτικό βίο και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις συμβάσεις που έχουν συναυθεί Επίσης, τι γίνεται με τα μικρότερα κρατημέλη. Πώς δεν θα μειονεκτήσουν σαν αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης. Ε, για όλα αυτά που ρωτήσατε, θέλω πάρα πολύ ώρα. Αλλά θα πρέπει να απαντήσω σε κάποια δευτερόλεπτα. Να, γιατί είπα, είναι ένα πρόβλημα το πώς όλα αυτά ε, συμβαδίζουμε τις ε, διατάξεις BEPS ε και του ΠΟΕ και για το εάν τα μέτρα που θα θεσπίσουν θα έχουν χαρακτήρα δεσμενούς διάκρισης. Όχι, δεν είναι αντίμετρα, δεν είναι αντίπεινα. Θα πρέπει για τις εταιρείε εκεί που γεννάται το κέρδος, εκεί να καταβάλλεται ο φόρος. Οπωσδήποτε να μην έχουμε διπλή φορολόγηση. Έτσι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο εταιρικό φόρο. Τώρα, όσον αφορά την πραγματική έδρα τη εταιρεία για τι ψηφιακέ εταιρείε, ε, αυτό καλύπτεται από το πνεύμα της πρότασή μα. Σήμερα έχουμε ως κριτήριο την πραγματική έδρα και ξέρουν πώς θα φορολογηθεί ένα τέτοιο εργοστάσιο, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις ψηφιακές εταιρείες. Ε, οπότε γι' αυτό και τώρα είπαμε να θα σπίσουμε μια σειρά κριτηρίων. Τη σύμβαση, το χρήστη κλπ. Αυτό, αυτό είναι το έργο που πρέπει να επιτελέσουμε. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Οι δε εταιρείε που αναφέρεται ακριβώς είναι εταιρείε που συλλέγουν δεδομένα. Αυτό γίνεται επί τη βάση και άρα εκεί θα πρέπει να κυριαρχήσει η διαφάνεια για το τα, τι δεδομένα χρησιμοποιούν και παρέχουν. Τώρα όσον αφορά τα όρια, τους περιορισμούς, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εταιρείε που ε, θα τα 750 εκατομμύρια ως τζίρο που πρέπει να φορολογηθεί και γι' αυτό και βάλαμε αυτό το όριο των 50 εκατομμύριων ευρώ για τις ε, εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ποστούν αυτή τη φορολογία. Γκίγκολτ, Σβέν. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε και πάλι στο βήμα αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας επενέσω για τα όσα κάνετε στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του εξαμήνου και των συστάσεων αναχώρα. Και είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν εύκολο να πείτε σε 7 κράτη-μέλη ότι πρέπει να αλλάξουν και να διαπιστώσετε ότι 9 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό για τις επιχειρήσεις. Θα με ενδιαφέρε αν μπορείτε να πείτε κάτι για το εάν θα δούμε Συστάσει ήδη τον Μάιο στι χώρες αυτές για να αλλάξουν την πολιτική του Επιπλέον θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή μα υπάρχει ένα νέο θέμα που ανακύπτει. Μιλάμε εδώ και καιρό για τον επιθετικό φορολογικό ανταγωνισμό όσον αφορά τις εταιρείε, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι όλο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός για το πού θα εγκατασταθούν τα πλούσια άτομα. Βλέπουμε κανόνες για τους ε, μη εγκατεστημένους ε, σε Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Κύπρο. Η Ιταλία έχει μια ειδική προσφορά για τα ξένα άτομα με μεγάλο πλούτο. Η Πορτογαλία δίνει μια δεκαετή φορολογική έκπτωση. Δηλαδή τα κρατημέλη ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν ε, πλούσια άτομα. Άλλη μια μορφή φορολογικού ανταγωνισμού μπορείτε να μας βοηθήσετε να ρίξετε λίγο φως σε αυτό το θέμα. Και στοχεύουν ε, και οι πίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν ξέρω αν ε, θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να αποκτήσουμε μια εικόνα για τα πλέον εκτίματα που υπόσχονται σε αυτά τα άτομα. Ελπίζω ως Ευρωπαίος Δημοκράτης που δεν κρύψατε ποτέ ότι ε, έχετε και σοσιαλιστικές ε, τάσεις να σας ενδιαφέρει το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Γκίγκολντ. Επιβεβαιώνω ότι η αντίδραση κάποιων υπουργών ε, των ΕΦΤΑ χωρών αυτών ήταν, θα έλεγα, αρκετά έντονη θα έλεγα κάπως διπλωματικά, όπως ήταν και η αντίδρασή μου. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν τους επιτεθήκαμε ως φορολογικούς ε, παραδείσους, όπως λένε κάποιες ΜΚΟ, γιατί έχουμε αυστηρούς ορισμούς, αλλά δεν έχει νόημα και να αρνούνται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οπωσδήποτε αυτός είναι ένας λόγος για να νομοθετήσουν. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω το εάν θα περιληφθούν αυτά στις ε, συστάσεις ε, ανά χώρα, γιατί ξέρετε ότι οι εκθέσεις αυτές αφορούν τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες και ελπίζω να γίνουν οι συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Με κάποιες υπάρχει ένα καλό πνεύμα διαλόγου, με κάποιες άλλες υπάρχει ακόμα άρνηση. Ελπίζουμε λοιπόν να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Για το υπόλοιπο σκέλος της ε, παραβασής σας, όχι μόνο ως ε, σοσιαλδημοκράτης, αλλά και ως ένας πολίτης ο οποίος επιθυμεί ισότητα και διαφάνεια και δικαιοσύνη, συμφωνώ με το πνεύμα των όσων είπατε, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο θέμα δικής μου αρμοδιότητας. Ε, αν δείτε παραδείγματος χάρη το πρόβλημα με τις χρυσές βίζες, σαφώς είναι αρμοδιότητας ε, της ε, συναδέλφου μου, της κυρίας Γιούροβα. Και ευχαριστώ να συνεργαστώ μαζί της. Αλλά ε, οι αρμοδιότητες μου δεν είναι τόσο περιορισμένες θα έλεγα, αλλά κυρίως αφορούν τους κανόνες για τις εταιρείε στην ενιαία αγορά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό το ζήτημα πράγματι. Και συμφωνώ και εγώ. Θα επανέλθουμε, λέει ο κύριος Γκίγκολντ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μαρή Πιερμπιέ. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Αχ, συγγνώμη. Κύριε Πίτροπε, πρώτα πρώτα μια παρατήρηση σε σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και την πολιτική κρίση που έχει χτυπήσει την Ευρώπη. Τώρα, ε, δεν μιλάμε ειδικολογικά, αλλά μιλάμε για κάτι ουσιαστικό, για τη μεταρρύθμιση πρώτα-πρώτα όσον αφορά αυτά τα, τα μέτρα, αυτό το 3% που είπατε, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 10% του φόρου του εταιρικού. Ο συντελεστής ο ζημινός, όπως είπατε, είναι 9,5% και σύμφωνα με την Επιτροπή είπαμε ότι από εδώ θα εκπέσει ο φόρος των εταιριών για να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση. Πρώτα πρώτα. Μα πώς θα παρακάμψουμε έναν ολόκληρο τομέα. Ο τομέα ο οποίος επειδή δεν έχει υλικό πραγματικό χαρακτήρα φοροδιαφεύγει. Και εγκαφά αυτά τα μέτρα πώς αυτά τα κούκκες δεν θα δεν θα μετακυλούνται στους καταναλωτές. Οπότε τώρα όσον αφορά πιο μακρόπνο μέτρα. Εδώ είναι το πρόβλημα ουσίας. Δηλαδή θα πρέπει να επανακαθορίσουμε το διεθνές φορολογικό δίκαιο και να δούμε τι θα γίνει με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς αυτό που είναι το 2017 τι μέτρα θα λάβουμε και η Ιρλανδία, οι κάτω χώρες, Κύπρος, Μάλτα, θα πρέπει να δούμε με τι στρατηγική θα σταματήσουν να φέρνουν την εμπλοκή. Γιατί η φορολογική παράδειση και η απάτη θεωρούμε ότι είναι δεσλειτουργίες όχι απλές λειτουργίες για την ΚΟΕ, αλλά είναι κάτι εγγενές μέσα στο ισχύον σύστημα και άρα θα πρέπει τα πράγματα να ανατραπούν. κοβίζει να ξεκινήσω από το τελευταίο που μας αναφέρατε. Μα αν θεωρείτε ότι τα χρηματοοικονομικά έχουν τα ενία της εξουσίας ή όχι, θα πρέπει βέβαια να γίνει το αντίστροφο. Γι' αυτό σας λέω ότι Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σε αυτό το πνεύμα κινούμαστε με ό,τι μέτρα να βάλουμε. Φυσικά και είναι διευθυντικού χαρακτήρα χωρίς να στερούνται της ηθικής πλευράς αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι μια πρόκληση στην οποία θα ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Τώρα όσον αφορά αυτό το οποίο μας είπατε για μακρόπνοα ή βραχυπρόθεσμα μέτρα. Ε, είπαμε ότι υπάρχουν λύσεις μακρόπνοες και βραχυπρόθεσμες. Γι' αυτό και προχωράμε με το άξιος όσον αφορά τις εταιρείε για το συντελεστή τώρα του 3%. Νομίζω ότι θα πρέπει να το θεωρήσετε αυτό που είναι, δηλαδή μια λύση. Λύση βραχυπρόθεσμη. Διαλέξαμε ένα τέτοιο συντελεστή. Θεωρούμε ότι είναι λογικός. Για δείτε. Πού οδηγεί ο Γκάφερ για αυτές τις ψηφιακές εταιρείες. Οι μισές αυτές τις εταιρείε είναι αμερικανικές, το εν τρίτον είναι ευρωπαϊκές και οι υπόλοιπες από τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι, δεν πρόκειται για δεσμένη διάκριση. Τους φορολογούμε τις δραστηριότητε τους. Πέντε δις ευρώ θα είναι το αρχικό έσοδο από αυτό το φόρο. Και επειδή αναπτύσσονται ταχύως αυτές οι εταιρείε, θα αυξηθεί και το έσοδο. Και να δούμε κατά πόσον θα θεωρηθεί αυτό το έσοδο μέρος των ιδίων πόρων. Και θα πρέπει ομόφωνα να αποφασίσει το Συμβούλιο. τελευταίο συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα με τέτοιο τρόπο που με κάνει αισιόδοξο ότι δηλαδή το Συμβούλιο θα υποστηρίξει την πρότασή μας αυτή. Και φυσικά θα προστατευτεί και ο καταναλωτής έναντι των μετεγκαταστάσεων. Γέζεκ. Να μην είστε εκτός θέματος συνάδελφοι, γιατί τη και θα έρθει ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης, Κόμπεν. Γεια σας. Κύριε Επίτροπε, εμείς δεν θέλουμε ότι είστε μόνο υπεύθυνο για τη βρολογία, αλλά είστε και λαμπρός υπουργό οικονομικών της Γαλλίας στο παρελθόν και ήρθατε σήμερα εδώ να συζητήσουμε τα φορολογικά και μας ε, αναφέρεστε βάσει της εμπειρία. της. Και τι θα έλεγε ένας υπουργός της Γαλλίας για κάποια τρίτη χώρα, ας πούμε, τη είπα και θα λέγατε ότι θα έχει ψηλότερη φορολογία η Γαλλία με κάποια συμφωνία που έχει γίνει. Και ότι όλα αυτά κάποιος επιδιαιτητής θα τα θεωρούσε παραβίαστη τη συμφωνία βουλευτή της Γαλλίας. Μα η απάντηση είναι ότι καμία χώρα δεν θα μπορούσε να συνάψει τέτοια εμπορική συμφωνία. Ούτε έχει γίνει αυτό ποτέ. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά έτσι να ταπεινωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω εδώ και αυτές τις guidelines, μας είπατε την Παρασκευή, ότι θα πρέπει η συμφωνία να οδηγήσει στο να σταματήσει ο προστατευτισμό του πλάσου Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, είπα, αυτά είπαν στον Ντέιβι. Και θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με Βασίλειο με τα πρόεδρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εφαρμογή ε, των μέτρων, αλλά θα υπάρχει και επιδιατησία ε, με αρμοδιότητα χρηματικών ποινών εις βάρος του Εμένου Βασιλείου. Μα τι είναι αυτό, αυτό είναι δικτατορία. Τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ή θέλει να οδηγήσει σε αδίέξοδο της προσπάθειας συμφωνίας. Πιστεύω ότι θα κάνω μια πολύ σύντομη απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, γιατί η ερώτησή σας ξεπερνάει το σημερινό μας θέμα. Ο κύριος Μπαρνιέ, ο οποίος διαπραγματεύεται εξ ονόματος των 27 κρατών μελών, όπως ξέρετε, φυσικά και όπως όλοι μας θέλει να φτάσει σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία να κρατήσουμε πολύ στενές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε την απόφαση να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει εν ευρωπαϊκή χώρα. Θέλουμε λοιπόν καλές συμφωνίες συνεργασίες μεταξύ ημών και θα το πετύχουμε. Τώρα, όσον αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία που έχουμε με την Βρετανική κυβέρνηση και όταν ήμουν υπουργό, αλλά και σήμερα σαν επίτροπος. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που στήριξε την ε, πρωτοβουλία του ΟΣΑ για την διάβρωση της φορολογικής βάσης, την ε, πρωτοβουλία BEPS και βεβαίως η Βρετανική κυβέρνηση στηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα για την δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων που βρίσκονται στον ψηφιακό τομέα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει φορολογικός παράδεισος. Φυσικά και θέλει να επιλέξει τη φορολογική του και την οικονομική του πολιτική και θα το κάνει και φυσικά και ε, θα έχουμε καλή συνεργασία μαζί τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται το, το οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με την φοροδιαφυγή και τώρα η ντράγκετα, η αγία, η μαφία ε, σε διεθνές επίπεδο αγοράζει, πουλάει εταιρείε, ομίλους συνοδοχείων κλπ. Και πολύ συχνά όπως είπατε και εσείς η Europol προσπαθεί να διευνήσει τι γίνεται με αυτά τα κρυπτικά νομίσματα. Επίσης άλλο θέμα. Είπαμε ότι έχουμε εκατομμύρια εμπορευομένων οι οποίοι έχουν ε, φτιάξει offshore εταιρείε που αντιστοιχούν σε δις ευρώ. Δεν υπάρχονται σε κάποιο έλεγχο όπως έχει σήμερα νομοθεσία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένω, δεν μπορούν να ανοιχνευτούν οι κινήσεις των ε, χρημάτων, των κερδών λόγω των φορολογικών παραδείσων. Και μια σειρά κυβερνήσεων στην Ιταλία έχουν ε, αντιμετωπίσει διάφορες ε, πολυεθνικές, τη Μισλέν, τη Φίλιπ Μόρις ε, και άλλες με τις οποίες να έχουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Μόνο το 2015 η Φίλιπ Μόρις στην Ιταλία έβγαλε κέρδη 1,33. Και βέβαια μέσω της Ελβετίας δεν καταβάλλονται σχετικοί φόροι και η Ευρώπη είναι αδρανής μάρτυρας όλων αυτών. Είναι σαφές, λέει ο Αυτά που μας λέτε είναι πολύ σημαντικά. Δεν αφορούν όμως μόνο το δικό μου χαρτοφυλάκιο της κυρίας Γιώργου και του Ντομπρόφσκης και άλλων συναδέλφων. Ναι, αναφέραμε για τα κρυπτονομίσματα σε σχέση με το πώς θα διέπονται από την νομοθεσία και αυτά τα σύστημα στο G20 να δούμε πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Οπότε και διατυπώσουμε αυτή μας την πρόταση για το πώς θα ρυθμιστεί η διακίνηση των μετρητών. Ε, βέβαια και θα πρέπει να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα μέσω του διασυνοριακού ΦΠΑ. Γιατί έχουμε τις φορολογικές απάτες με το ΦΠΑ που κοστίζει στα κρατημέλη 50 δις. Και πού πάνε αυτά. Ναι. Πολύ συχνά ε, χρηματοδοτούν το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία. Άρα, για να προχωρήσουμε την πρότασή μας, θα πρέπει ο ΦΠΑ διασυνοριακός να έχει την ίδια ρύθμιση όπως και ο ΦΠΑ σε κάθε χώρα. Έτσι θα τους αντιμετωπίσουμε αυτού τους εγκληματίες. Και το Συμβούλιο γι' αυτό κατήρτισε την μαύρη λίστα για τους φορολογικούς παράδεισους ούτως ώστε να βρεθεί κάποια λύση και να υιοθετηθούν κάποια πρότυπα καλής διακυβέρνησης να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια στον νόμο. Ποιος μπορεί και έτσι ζητεί να δευτερολογήσει. Όχι, όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος. Γιέζεκ. Α, του δίνει το λόγο. Όχι. Ο Γιέζεκ είπε όλοι έχουν τοποθετηθεί και έχουμε σύμφωνα με το κανόνα του Ντόν τέσσερις αγορητές. Ε, και πρώτα πρώτα για το ΕΛΚ, Νίντεμάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Επιτροπέ. Η πρώτη ερώτηση αφορά την ψηφιακή φορολογία. Το πρώτο θέμα είναι αν υπάρχει κάποια συζήτηση των αρχών μέσα για το πώς θεωρούν το ότι πώς βλέπουν ότι κάποιες εταιρείε ε, έχουν κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να φορολογούνται εδώ. Δεύτερον, για την εφαρμογή αυτή του οποίου λέτε θα χρειάζεται και συνεργασία των εταιριών για να έχετε τα δεδομένα επί τη βάση των οποίων θα υπολογιστεί ο φόρος. Πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο. Και μετά είχα μια παρόμοια ερώτηση προς τον κύριο Αλένα Μασόρ για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, αλλά Βλέπω από την απάντησή σας ότι είναι απίθανο η Βουλγαρική και η Αυστριακή Προεδρία να πετύχουν ε, κάτι αν σκεφτούμε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις υψηλού επίπεδου και πολλές χώρες είναι εναντίον. Οπότε σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητο να πάμε προς μια ενισχυμένη συνεργασία για να πετύχουμε τουλάχιστον κάτι. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα μετά από αυτό το οποίο είπε και ο Ρομπέρτο Παλτιέρη ότι ε, συμφωνώ ότι ε, καλύτερο τρόπο είναι να φορολογήσουμε τα κέρδη και όχι τον τζίρο. Γι' αυτό νομίζω ότι η βραχυπρόθεσμη λύση είναι ακριβώ αυτό, βραχυπρόθεσμη. Δεύτερον, για τα δεδομένα. Όπω όλοι σχεδόν οι φόροι στι εταιρείε θα είναι κατά δήλωση ε, πως γίνεται και για τα άτομα. Θα πρέπει να δώσουν λοιπόν τα δεδομένα. Όλες οι επιχειρήσεις τις οποίες ε, συνάντησα μου είπαν ότι θα συμμορφωθούν με τους κανόνες. Οπότε σε εμά επαφίεται να διαμορφώσουμε τους κανόνες. Εάν οι κανόνες ε, απαιτούν ότι θα δηλώσουν ε, τι κάνουν με τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Όσον αφορά την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ποτέ δεν ξεχνάω τα τρία σε. Αν και θα δεχόμουν μια προσέγγιση δύο φάσεων, αλλά θα πρέπει να τις, να τις δούμε πάντα ως σύνολο. Πρέπει να αποφασιστούν αυτά μαζί και ταυτόχρονα. Και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό. Και το δεύτερο, για την ενισχυμένη συνεργασία πλέον δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια προσπάθησα πρώτα απ' όλα ως Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και μετά ως Επίτροπος για να πιέσω κάποια κρατημένη να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ε, και όπως βλέπετε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο παρά μόνο τώρα οπότε δεν σημαίνει ότι είναι απλούστερο το να προχωρήσουμε σε ενισχυμένη συνεργασία, το να συμφωνήσουν 28 και αύριο 27 και νομίζω ότι θα εγκριθεί τελικά η κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων πριν το τέλος του έτους. Σοσιαλδημοκράτης, κυρία Βερές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μας είπατε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη της ΤΑΚΣΤΡΙΑ 3 και η ολοκλήρωση των προσπαθειών μεταρρυθμίσεων. Μπορείτε να μας πείτε όμως Πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί αν δεν έχουμε ακόμα τις τελικές σας προτάσεις και πώς ε, θα μας βοηθήσετε και εσείς να περάσουμε προς το τελικό σύστημα από το προσωρινό και την προσωρινή σειρά μέτων που προτείνεται σήμερα. Όσον αφορά τους εταίρους μας, τους Αμερικανούς, οι οποίοι μιλούν για κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης ε, στον κόσμο της ψηφιακής οικονομίας. Η πρόταση CCCTB βεβαίως δεν στοχεύει μόνο τον κόσμο της ψηφιακής οικονομίας, αλλά τον σύνολο των πολυεθνικών που σήμερα φορο... χρησιμοποιούν τεχνικές φοροαποφυγής. Τέλος, θα ήθελα να σας καλέσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να είναι σε μια φάση αναδιάρθρωσης, ανασχηματισμού της πολιτικής της σκέψης. Μήπως θα μπορούσατε να ξεκαθαρίσετε λίγο και να αποφασισαφηνίσετε τις ε, τεχνικές ε, που αφορούν την ε, νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες διαδικασίες, τη λεύκαση χρήματος δηλαδή. Ε, ίσως, και θα μου πείτε ότι είναι αρμοδιότητες της κυρίας Γιούροβα, ίσως αυτή η μονάδα λεύκανσης βρώμικου χρήματος θα πρέπει να ενσωματωθεί στις δικές σας αρμοδιότητες. Ευχαριστώ κυρία Πέρεστα. θα απαντήσω στις τρεις ερωτήσεις σας. Πρώτον, οι προτάσεις για το ΦΠΑ φυσικά και θα συμπληρωθούν και αυτό το Μάιο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με έναν πιο ολοκληρωμένο και πλήρη τρόπο. Όσον αφορά το CCCTB, την ενοποιημένη κοινή βάση για την φορολόγηση των εταιριών, Κοιτάξτε, εκεί πραγματικά για μένα βρίσκεται και ο ακρογωνιαίος λίθος για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας για τον 21ο αιώνα. Όμως δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη στο να υιοθετήσουν σε μια πρώτη φάση την προσωρινή ε, μεταρρύθμιση και πρότασή μας. Δεν ξέρω, και τώρα πάω στην τρίτη σας ερώτηση, αν βρισκόμαστε σε μια φάση σκέψης για την αναδιάρθρωσή μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως όταν ανανεωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, θα πρέπει να κάνετε αυτή την ερώτηση στον διάδοχό μου. Το ΕΛΚΟ, Μπράιν Χέιζ, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Τρεις ερωτήσει Πρώτα απ' όλα, μια πολιτική ερώτηση. Δικαίω λέτε ότι οι μισές εταιρείε που επηρεάζονται από την ενδιάμεση αυτή η πρόταση είναι αμερικανικές. Αν ισχύετε για μια ανταπόδοση από τις ΕΠΑ, καθώς μιλάμε ε, για μια κυβέρνηση η οποία είναι η πιο προστατευτική που έχουμε δει σε θέματα διεθνούς εμπορίου στις ΗΠΑ. Η δεύτερη μου ερώτηση, μιλάτε τώρα για μια λύση μέχρι το 2020 με μια ενημερωμένη πρόταση από το 2019 ε, βλέπετε κάποια πιθανότητα να αντιδράσει πιο γρήγορα ο ΣΑ στο θέμα αυτό της ψηφιακής φορολογίας, όπου συμφωνώ ότι το ποσοστό είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο περιμέναμε και πρέπει να το δούμε. Τελευταία μου ερώτηση. Βλέπετε την ε, δυνατότητα σταδιακής κατάργησης ε, της πρότασής σας μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση στο επίπεδο του ΟΣΑ θα δούμε βέβαια και θα γίνει με την κοινή φορολογική αίλη των επιχειρήσεων αναλόγω με την στήριξη που θα βρει. Αλλά μήπω θα μπορούσαμε να προωθήσουμε γρηγορότερα την ε, πρόταση του ΩΣΑ και μετά να ακολουθήσει και η δική σας η πρόταση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές που είναι πραγματικά θεμητές. Θα ξεκινήσω με τον ΩΣΑ. Εκτιμώ την δουλειά που γίνεται εκεί και θεωρώ ότι η έκθεση αυτή του ΩΣΑ πριν από 15 μέρες είναι υψηλής ε, ποιότητας. Ε, τι μας λέει. Μας δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ότι δεν υπάρχει συνένεση και ότι πρέπει να εργαστούμε για να οικοδομηθεί η συνένεση μετά το 2020 και δεν μπορούμε νομίζω να σπαταλήσουμε τόσο χρόνο. Και βλέπω τώρα κάποια κράτη-μέλη ε, θεωρούν ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να νομοθετήσουν από μόνα τους. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά μόνοι μας και γρήγορα. Η ενδιάμεση λύση εξορισμού ε, θα πρέπει να είναι ενδιάμεση. Όχι μόνο ένα αναμονή τη κοινή φορολογική βάσης των επιχειρήσεων, αλλά αναμένοντας μια συνολική προσέγγιση του ΩΣΑ και των νομικό ορισμό της ψηφιακής παρουσίας ε, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί βεβαίω ε, ιδανικά στην κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων ή σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος, για την αντίδραση των ΙΠΑ, όπως ξέρετε, έχω απευθύνει μια επιστολή στον Στίβεν Μενούτσι, τον Υπουργό Οικονομικών, ε, τον συνάντησα και στο Μπουένος Άιρες, είχα την ευκαιρία να του μιλήσω στην συνάντηση των ε, G20 και παραλαμβάνω εδώ ότι πρώτον ο φόρος τον οποίο ε, προτείνουμε δεν στρέφεται κατά τον ΙΠΑ, είναι κάτι το οποίο κάνουμε εμείς, ε, το οποίο μας απασχολούσε εδώ και μήνες και δεν είναι αντίδραση σε εμπορικέ κινήσεις που νομίζω ότι είναι πλαπτικές, αλλά δεν στρέφεται κατά τον ΙΠΑ γιατί οι εν λόγω εταιρείε δεν είναι καθόλου αμερικανικές, κάποιες είναι, κάποιες άλλες εξαιρούνται και δεν είναι φόρος για Google, Amazon, Facebook ε, κτλ. Ε, είναι εντυπωσιακό βεβαίως γιατί ο κόσμος είναι μαθημένος ε, να ακούει για αυτές τις εταιρείε, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αφορά γύρω στις 80 εταιρείε που καλύπτονται από αυτόν τον φόρο. Και αυτό θα πω και όταν θα μιλήσω στους Αμερικανούς φίλους μας στην Ουάσιγκτον σε λίγες εβδομάδες στην συνέλευση του Δέλτα Και θα τα πω και στον Λευκό Οίκο, στο Υπουργείο των Οικονομικών, για να μην υπάρξει έτσι μεγάλη αναστάτωση. Σας ευχαριστώ. Πολ Τάγκ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις κύριε Μοσκοβισή. Έχουμε τις ίδιες απόψεις, αλλά όταν παρουσιάσατε το ψηφιακό πακέτο αναφερθήκατε στους ε, γίγαντες τεχνολογίες που πληρώνουν 9% ε, ε, κατά μέσο όρο φόρο. Αλλά είναι αρκετά ψηλό θα έλεγα. Η Apple σύμφωνα με την Κομισιόν πλέον 0,05% και έχω δει ότι η Google ε, πλήρωσε 46 εκατομμύρια το 2016 ε, με ε, επιτζήρο 22. Μήπως θα μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τον φόρο που πληρώνουν αυτοί οι γίγαντες ή δεν πληρώνουν. Δεύτερη ερώτηση. Η συνεργασία με τις χώρες. Ήμουν χτες στην Ολλανδική Βουλή, βλέπω ότι τα μελετάει ακόμα η Ολλανδική κυβέρνηση. Ε, χρειάζεστε την συνεργασία των κρατών μελών για να υπάρξει ακριβώς ε, ε, μια μελέτη αντικτύπου για τον ψηφιακό φόρο στις χώρες αυτές και μπορείτε να μας πείτε εδώ στο Κοινοβούλιο ποιες χώρες και ποιες φορολογικές διοικήσεις δεν συνεργάζονται για να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται στις χώρες και σε σχέση με αυτό, ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 116 και θα πέρασει σε ειδική πλειοψηφία. Γιατί να μην περιλάβετε και αυτό το άρθρο σε αυτό το πακέτο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έδωσα δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε στοιχεία εθνικά, για την κάθε χώρα δηλαδή και για την κάθε επιχείρηση στην κάθε χώρα. Φυσικά και θα πρέπει και βάσει της εργασίας της συναδέλφου Επιτρόπου να βρούμε πού υπάρχουν τα αδύναμα σημεία, οι αδύναμοι κρίκοι, τους οποίους φυσικά χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να φοροαποφύγουν. Και χρειάζεται εδώ να συνεργαστούμε όλοι, να ανταλλάξουμε στοιχεία, έτσι ώστε να υπάρξει μια δίκαιη φορολόγηση στα σωστά επίπεδα που ανταποκρίνονται στα πραγματικά τους κέρδη. Και φυσικά και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις, με τα εθνικά κοινοβούλια, για να υπάρξει και βελτίωση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τον επιθετικό ορολογικό σχεδιασμό. Ένιωσα και όταν είχα επαφή με τον ε, κύριο Μέλ στις κάτω χώρες ότι υπήρξε μια σχετική ανταπόκριση, βελτίωση της αντίστοιχης νομοθεσίας. Εγώ δεν ένιωσα αυτό που μου περιγράφεται, ένα πλήρες, μια πλήρη άρνηση. Φυσικά πάντως η εργασία μας με τα κράτη-μέλη είναι κάτι που μας απασχολεί και θα το συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας εδώ στην ανταλλαγή απόψεων και στη συζήτησή μας. Αυτή η συζήτηση μας δείχνει με σαφήνεια ότι έχουμε mm. τους ήχους τους ίδιους στόχους όσον αφορά τη φορολογία, όσον αφορά τη φορολογική μας στρατηγική και όλοι προσβλέπουμε να υιοθετηθεί ένα σύστημα με μία δίκαιη φορολογία. Θέλω να διευκρινίσω mm. κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπήρξε διαδικασία catch the eye έδωσα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής βάσει μιας προκαθορισμένης λίστας. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τη δέσμευσή του, για τις προσπάθειές του. Είμαστε, όπως είπατε, όλοι σε αυτόν τον κοινό αγώνα, αποφασισμένοι και δεσμευμένοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να πιέσουμε, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε για να υιοθετηθούν τα μέτρα αυτά από αυτό το Κοινοβούλιο και από αυτήν την Επιτροπή. Κάναμε ένα καθοριστικό βήμα μπροστά, ένα καθοριστικό βήμα πρόοδου. Κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την συνολική στρατηγική αυτής της Επιτροπής. Και ο ρόλος σας είναι καθοριστικός, κύριε Επίτροπε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επιτέλους εργαλεία και μέσα για να υπάρξει μια δίκαιη φορολογία που να ισχύει σε όλους τους τομείς και εδώ ιδιαίτερα μας αφορά ο τομέας ο ψηφιακός και οι μεγάλες πολυεθνικές. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία επιτρέπει σε κάποιους να ξεφεύγουν. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ευχαριστώ.